συνέταξη με την έκθεση του κυρίου Κάριμ, ετήσει εκθέσεις 2012-2013 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Καρίμ να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλό απόγευμα σε όλους ένας συνάδελφος με χιούμορ μου είπε προηγουμένως προσβλέπω ιδιαίτερα στις ετήσιες προτάσεις σας για την ε, ε, αναλογικότητα και την επικουρικότητα. Και εγώ απλώς χαμογέλασα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα πολλά χρόνια που μπορώ να παίξω και εγώ κάποιο ρόλο για να μπορέσω να διαμορφώσω τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζεται η διαδικασία νομοθεσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά δεν μπορώ να το αλλάξω μόνος μου και γι' αυτό θα πρέπει να εκφράσω την τις ευχαριστίες μου σε όλους τους τις συζητές, οι οποίοι ο Σουεύκα, η κυρία Χόφμαν, ο Πιν, Μαρίνο Ιππίντο, όλοι αυτοί οι συνάδελφοι όπως και η Αγγέλικα Νίμπλερ η οποία φεύγει τώρα από την Ολομέλεια ενώ αναφέρομαι σε αυτήν που με βοήθησαν πάρα πολύ. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη χώρα μου το Ενωμένο Βασίλειο. Εγώ πιστεύω <clears throat> πράγματι ότι η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο ισχυρές και οι δύο όταν βρίσκονται μαζί και μέσα από τις προτάσεις μας μπορούμε να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ αυτού του Κοινοβουλίου και του Εθνικού Κοινοβουλίου στην Μεγάλη Βρετανία. Η συμμετοχή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βοηθήσει και έχει ενισχύσει το σύνολο της Ευρώπης. Αλλά ίσως αυτή είναι μία από τις τελευταίες ευκαιρίες που εγώ ως Ευρωβουλευτής έχω τη δυνατότητα να θέσω προτάσεις όπως αυτές που θα σας παρουσιάσω γιατί θα ακολουθήσει το δημοψήφισμα για την παρουσία της, μεγάλη βρετανία Μεγάλης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ιδιαίτερα αμφίροπο. Τι είναι λοιπόν αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες μας για το θέμα αυτό. Μπορεί να μην αναγνωρίσουν τις λεπτομέρειες και τα ονόματα που δίνουμε στα θέματα αυτά, αλλά πολύ συχνά μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ απόμακρη. Κάνει πάρα πολλά πράγματα και αυτά που κάνει επηρεάζουν χωρίς λόγο και αρνητικά πάρα πολλούς ανθρώπους. Εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτά τα κομβικά θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη δική μας τη δημοκρατική λογοδοσία. Ιδίω αν αυτές οι μεταρρυθμίσεις απορρίπτονται, εμείς ουσιαστικά βοηθάμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να διασπάσουν και να κατακαιρματίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποδυναμώσουν τους πολίτες μας. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν οι ηγέτες μας έφτασαν σε μία συμφωνία και έχουν υποβάλει σε μας αυτήν την συμφωνία να δούμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απόμακρη η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και τα δικαιώματά τους και οι υποχρεώσεις τους θα πρέπει να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν περισσότερο στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης απόφασης μόνο. Έτσι ενισχύουμε τα κοινοβούλια αυτά και τους εαυτούς μας. Πρέπει να αποδεχτώ ότι η δική μας Επιτροπή Ελέγχου για τα Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βουλή των Κοινοτήτων δεν είναι ιδανική και δεν θέλω να την παρουσιάσω ως υπόδειγμα αν <clears throat> επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να έχουμε την Ευρώπη μόνο όταν τη χρειαζόμαστε. Αυτό είναι η επικουρικότητα. Έχουν αυξηθεί οι θέσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων στην νομοθεσία, αλλά δεν συμμετέχουν όλα τα κοινοβούλια. Και όπως λένε και οι διάφορες μελέτες, δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς η επικουρικότητα στις εκθέσεις αντικτύπου μας. Εγώ πάντα λέω ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στην εκπόνηση τη νομοθεσία, όπω είναι οι λευκές βίβλοι και οι πράσινε βίβλοι. Μπορεί να υπάρχουν και αιτήσεις επαφέ και συναντήσει των Εθνικών Κοινοβούλων Κοινοβουλίων με την Κομισιόν. Η διαδικασία της κίτρινης κάρτας θα πρέπει να εφαρμόζεται με ευκολία στα εθνικά κοινοβούλια. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες για αυτή τη διαδικασία. Και θα πρέπει να παραταθεί το διάστημα 8 εβδομάδων για τον έλεγχο επικουρικότητας των 8 εβδομάδων. Είναι λοιπόν πολλές προτάσεις, τις οποίες δεν θα τις αναφέρω επακριβώς, αλλά όταν επανέλθω στο τέλος της συζήτησης θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι η τελική μου έκκληση είναι εξή. Δεν πρέπει να φοβηθούμε όταν λέμε ότι πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας και τα εθνικά κοινοβούλια μεγαλύτερη δυνατότητα να συνεργαστούν ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να καταλήξουμε σε νομοθεσία η οποία έχει σχέση με τους πολίτες μας και τους βοηθά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την εξαιρετική σας έκθεση που αφορά το 2012-2013, επικουρικότητα και αναλογικότητα. Για την Επιτροπή Αναλογικότητα και Επικουρικότητα θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σαφώς και είναι ένας από τους στόχους μας για όλες τις πολιτικές μεγάλες και μικρές. Έχουμε δεσμευθεί ότι η αρχή της επικουρικότητας θα υπάρξει σαν πραγματική διαδικασία από όλους τους θεσμούς έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη δράση, καλύτερη κατανόηση έτσι ώστε κάθε πρόταση που αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική να λαμβάνει υπόψη της αυτήν την αρχή. Κάθε φορά που καλούμεθα να παρακολουθήσουμε, να ελέγξουμε το σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, εμβαθύνουμε τη σχέση μας με τα εθνικά κοινοβούλια όταν αυτό γίνεται εγκαίρος στα εθνικά κοινοβούλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει λοιπόν νέες σχέσεις, νέες εταιρικές σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια, με πολύ πιο συχνές επισκέψεις της Επιτροπής στα Εθνικά Κοινοβούλια. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2014 η επίτροποι έκαναν πάνω από 270 επισκέψεις στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να αυξάνουμε την συχνότητα αυτών των επισκέψεων, των επαφών, για να εξηγήσουμε καλύτερα τι κάνουμε και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να δώσουμε απαντήσεις στις ανησυχίες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όλα αυτά βεβαίως και βάσει της διαδικασίας για την μελέτη αντικτύπου. Όπως ξέρετε το 2014 και 2015 υπάρχει μια σειρά νέων μέτρων για τον καλύτερο, την καλύτερη αξιολόγηση αντικτύπου, περισσότερη διαφάνεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενισχύσει και τις μελέτες αντικτύπου και τις αξιολογίες αντικτύπου αλλά και τις αποστεριόρι αξιολογήσεις, βασιζόμενοι πάντα σε μία ανάλυση της αναλογικότητας και της χρήσης επικουρικότητας. Οι πτυχές λοιπόν της επικουρικότητας και της αναλογικότητας είναι πάντα στην καρδιά αυτής της αξιολόγητης, είτε γίνεται εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων. Και Σκοπός μας είναι να κάνουμε συστάσεις για βελτίωση της ισχύω της αρχής της επικουρικότητας και να εξετάζουμε κάθε φορά αν η αναλογικότητα και η επικουρικότητα έχουν ληφθεί υπόψη. Αυτό ζητείται από όλους τους θεσμούς έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η επικουρικότητα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη πριν υιοθετηθεί ένα κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη γιατί τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν στην διοργανική τους συμφωνία την καλύτερη νομοθεσία με επίκεντρο την αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας που θα πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση όταν προετοιμάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και ο αντίκτυπός της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε περίπτωση προτείνει συγκεκριμένα μέτρα καθώς και την υλοποίησή τους βάσει της αρχής της αναλογικότητας και της υπηκότητας και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κάνει αξιολογήσεις αντικτύπου προτείνοντας πολύ συγκεκριμένες τροπολογίες και υποβάλλοντάς τις ε, στις αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα τρία θεσμικά όργανα έχουν δεσμευθεί και θεωρούν ότι η επικουρικότητα είναι ένα καθοριστικό στοιχείο της όλης νομοθετικής διαδικασίας. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε η επικουρικότητα και η αναλογικότητα να παραμείνουν στην καρδιά της δημοκρατικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάσει της ε, διοργανικής ε, συμφωνίας πλαισίου θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να γίνεται σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιαστόφσκι έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Καρύμ για αυτήν την έκθεση. Για το αναλυτικό κομμάτι, αλλά και για το κομμάτι που περιλαμβάνει και προτείνει μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως, πρόκειται για μια ε, έκθεση εξαιρετικά βρετανικού τύπου. Δηλαδή, ε, εφόσον πούμε ένα α, θα πρέπει να πούμε και το β. Ε, δηλαδή θα πρέπει να αποκομίσουμε ε, τα συμπεράσματα και να αναλάβουμε τις επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά για αρχές αναλογικότητας και επικουρικότητας και θα πρέπει και η ίδια να είναι πιο συνεπής. Αυτές οι έννοιες δεν είναι αφηρημένες ή επικουρικότητα συνδέεται με το ορθό δίκαιο, την ορθή νομοθεσία, χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία, χωρίς ε, δυσκολίες για τα κράτη-μέλη. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, δηλαδή να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε σε σχέση με τις δυνατότητες των κοινοβουλίων να χρησιμοποιήσουν την επικουρικότητα ε, και είμαι πεπισμένος και θέλω το, Ευρωπαϊκό, το Ηνωμένο Βασίλειο να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και για να, να σκεφτούμε και το κόκκινη κάρτα για να μπλοκάρουμε μια κακή νομοθεσία να είναι ενιαία κριτήρια που θα οργανώνουν τη συνεργασία ανάμεσα στα κοινοβούλια και τα κράτη-μέλη. Περισσότερο άνοιγμα, περισσότερο θάρρος από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πρέπει να μην αντιμετωπίζει τα εθνικά κοινοβούλια ως ανταγωνιστές όπως είπε και ο εισηγητής. Ελπίζω και πιστεύω πως και το Ηνωμένο Βασίλειο θα μείνει εντός Ένωσης γιατί η συμβολή του είναι θετική για τη σωστή ορθή νομοθεσία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο, η κυρία Στίβενς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ως εισηγητής γνωμοδότηση στην Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη γιατί πολλά από τα στοιχεία τη γνωμοδότησή μα περιλήφθηκαν στην έκθεση του κυρίου Κάριμ στην Νομική Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από συστάσει. Θέλουμε πρώτα απ' όλα η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να συζητήσουμε περισσότερο για την εφαρμογή τη αρχή τη αναλογικότητα και της επικουρικότητας στα κοινωνικά θέματα. Δεύτερον, για τα θέματα της ε, επικορικότητας θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια προσθέμενη αξία. Εγώ συμφωνώ επίση και με μερικές ανησυχίες που εκφράστηκαν. Θα πρέπει οι εκθέσεις αντικτύπου να γίνονται από μια ανεξάρτητη αρχή. Νομίζω λοιπόν να υπάρξουν οι απαραίτητες τροποποίησεις για την νομοθετική διαδικασία στην πρόταση της Πρέπει να δούμε επίση κατά πόσο οι τροπολογίε οι οποίε ε, εφαρμόζονται σε μια έκθεση ανταποκρίνονται στην αρχή τη επικουρικότητα. Κύριε Σούλιν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καρίμ για την έκθεση την οποία έχει προετοιμάσει. Εγώ χαίρομαι ότι οι προτάσεις του είναι όλες προτάσεις που εμείς έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εάν ακολουθήσουμε τις αρχές της και της αναλογικότητας, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια νομοθεσία η οποία θα είναι προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Εμείς έχουμε κάνει πάντα προσπάθειες η Κομισιόν να μπορεί να κάνει αυτές τις ε, πολιτικές για να είναι αποτελεσματική η δράση Η Κομισιόν θα πρέπει να καταδείξει με καλύτερο τρόπο πού είναι η προσθέμενη αξία των προγραμμάτων και να σχεδιάζει καλύτερα τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές. Θα πρέπει να γίνεται η έκθεση για την επικουρικότητα κάθε πρότασης και να αποδεικνύεται ότι πράγματι ισχύει αυτό. Η κυρία Μπεγκίν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ παρεμβαίνω εξ ονόματο του Ντάβιτ Μπορέλη, που είναι εισηγητή για γνωμοδότηση τη Επιτροπή ΙΝΤΑ. Το θέμα τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα είναι κεντρική σημασία για την αρμονική ανάπτυξη των νομοθετήτων τη κοινότητα, γιατί αφορά τη συνεργασία ανάμεσα στου πολίτε και τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, δεν αναφέρεται στην πολιτική την ε, συγγνώμη, επηρεάζει και την εμπορική πολιτική και γι' αυτό ήθελα να συνοψίσω τη συζήτηση που κάναμε στην ΙΝΤΑ. Πρώτα απ' όλα έχουμε το θέμα των ε, ISDS, των ε, διαιτησιών ανάμεσα... Ο πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια, παρακαλώ, μιλήστε λίγο πιο αργά. Πρώτα απ' όλα έχουμε λοιπόν τις διατησίες, κατά δεύτερο λόγο έχουμε την μακροοικονομική βοήθεια, περισσότερους εκ των προτέρων ελέγχους και εκ των υστέρων και ιδιαίτερα για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την αναλογία της βοήθειας που προσφέρουμε στους εταίρους μας, ενώ θα ενισχύσουμε τον έλεγχο τον κοινοβουλευτικό. Κατά τρίτο λόγο υπάρχουν τα θέματα της διαφάνειας και των αξιολογήσεων αντικτύπου των διεθνών ε, συμβάσεων και συνθήκων. Η εμπλοκή των εταιριών σε αυτή τη φάση και κυρίως των μικρομεσαίων είναι ε, απαραίτητη. Για, τέλος, ε, θα θυμίσω την, αλληλεγγύη και, την επικορικότητα και την αναλογικότητα ως κεντρικό ζήτημα των εμπορικών μας ε, συζητήσεων. Θα πρέπει να θεωρήσουμε πως η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να αποκλειστεί από αυτό το πλαίσιο επικορικότητας και αναλογικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Σβίφκα, δύο λεφτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και πολλά χρόνια μιλάμε και ε, συνεργαζόμαστε με μεγάλη χαρά με τον εισηγητή για αυτό το ε, σημαντικό θέμα. για αυτά τα θέματα της, αλληλεγγύ... της ε, αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Ε, κάθε φορά εγκρίνουμε νέες προτάσεις και προβαίνουμε σε βάθος αναλύσεις για το τι πρέπει να κάνουμε. Καλό... Θα άξιζε τον κόπο να προβούμε σε συγκεκριμένες δράσεις γιατί αμφίβολα αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του δικαίου. Η αναλογικότητα και η επικουρικότητα είναι θεμελιώδη σημασία στο νομοθετικό πλαίσιο και την νομοθετική διαδικασία της Ένωσης. Θα έλεγα ότι το σημείο εκκίνησης ε, μάλιστα είναι για το κοινοτικό δίκαιο. Κυρίως εφόσον στα κρατημέλη <coughs> βλέπουμε να αυξάνονται οι φωνές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, γιατί ε, βασιζόμενοι στην ε, περίπλοκη νομοθεσία Γι' αυτό και με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα μαζί με μια διαδικασία αξιολόγησης ε, των επιπτώσεων των νομοθεσιών ε, θα ήταν θεμελιώδη σημασία. Θα πρέπει δηλαδή να συνδέσουμε τις δραστηριότητές μας με την ε, αντίληψη περί του δικαίου όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Να καταλάβουν δηλαδή γιατί έχει προστιθέμενη εξή ευρωπαϊκή νομοθεσία και ότι δεν είναι κάτι το οποίο το προτείνουμε έτσι, ε, ειδικά τα, ευρωπαϊκά, τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερα στην εκπόνηση και στην σύνταξη νέων νομοθεσιών. Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε ώστε στην έκφραση της γνώμης τους να συμμετέχουν, να είναι πιο δραστήριοι. Αυτό αφορά τόσο τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και το τελικό ε, δίκαιο, τις τελικές νομοθεσίες που θα προκύψει ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θεωρώ πως οι προθεσμίες για την υποβολή των θέσεων των, των Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει να παραταθούν. Να ενισχυθεί δηλαδή ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η πρόταση δηλαδή του εισηγητή να εισαχθεί αυτή τη πράσινη κάρτα που θα επέτρεπε στα εθνικά κοινοβούλια να υποβάλουν λογικές και βάσιμες προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, πιστεύω πως είναι μια πολύ θετική πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντελβό, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε ποιο βαθμό οι αρχές αναλογικότητας και της επικουρικότητας είναι πολύ σημαντικό για να δημιουργήσουμε μια Ένωση Ευρωπαίων Πολιτών. Χρήσιμες αρχές για την καλή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στην καλή λειτουργία. Σε καμία περίπτωση αυτές οι αρχές δεν έχουν σκοπό να μην λειτουργήσει αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας θα πρέπει να εξισορροπούνται από την ορθή και αποτελεσματική ε, λειτουργία των θεσμών μας. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ισορροπία. Θεωρώ ότι η έκθεση όπως παρουσιάζεται τελικά απειλεί αυτήν την πολύ λεπτή ισορροπία και την ορθή λειτουργία θα ήθελα πραγματικά να δημιουργήσουμε αυτές τις ε, προϋποθέσεις έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε το κλίμα του ευρωσκεπτικισμού που επικρατεί στην Ευρώπη. Να ενισχύσουμε την νομοθετική διαδικασία και να μην βαρύνουμε την γραφειοκρατία η οποία ήδη υπάρχει και παρεμποδίζει την ορθή λειτουργία των θεσμών μας. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία. Οφείλουμε όμως τους πολίτες μας μια αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες τους, μια αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ευέλικτη Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να φέρνει πιο κοντά τους λαούς οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις κοινέ προκλήσεις. Εξ λοιπόν αυτών που πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώ όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τις τροπολογίες της ε, ομάδας μας, της ομάδας των σοσιαλδημοκρατών για την στήριξη αυτής της αρχής της αναλογικότητας και της επικουρικότητας στήριξη αλλά όχι δίνοντας περισσότερη ανισορροπία. Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ με την θέση του εισηγητή όσον αφορά την αναλογικότητα και την επικουρικότητα. Τον ευχαριστώ όμως για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Ένα λεπτό κυρία Χένκελ. Θέλω να ευχαριστήσω την, τον κύριο Καρύμ στα γερμανικά βέβαια δεν υπάρχει άλλη χωριστή λέξη για την επικουρικότητα από το subsidiarity. Τι σημαίνει αυτό. Αν έχουμε ένα πρόβλημα στο Αμβούργο πρέπει να το λύσουν οι Χαμβουργέζοι. Και όχι να προσπαθήσουμε να το φέρουμε στο Βερολίνο. Αν δεν μπορεί να λυθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο στι Βρυξέλλε, μόνο τότε θα πρέπει να έρθει στι Βρυξέλλε. Αλλά εδώ γίνεται πάντα το αντίθετο. Παραβιάζεται η αρχή τη επικουρικότητα γιατί θέλουμε να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση της Ευρώπης, κάτι το οποίο οδηγεί νομοτελειακά σε μια συγκεντρωτικότητα. Αυτό απομακρύνει περισσότερο τους Ευρωπαίους από τις Βρυξέλλες και την Ευρώπη, οδηγεί σε μια ελίπουσα ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης και στην ανάδυση των ε, ακροδεξιών και ριζοσπαστικών απόψεων. Θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε να καταλάβουμε ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτή την συγκεντρωτική διαδικασία που οδηγεί μόνο σε περισσότερη συγκέντρωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρίνιου Ιππίντου, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω το έργο του εισηγητή που ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με την έκθεση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η απόσταση που νιώθουν οι πολίτες και κάποια κράτη-μέλη από τους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι η έκθεση του κυρίου Καρύμ ξεκινά από αυτή την αφετηρία, από αυτή τη διάγνωση και προσπαθεί με αυστηρότητα και με σοβαρότητα να κατανοήσει πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της αναλογικότητος και της επικουρικότητας. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να δώσει περισσότερη ε, στεναρότητα στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρει τους θεσμούς αυτούς πιο κοντά στους πολίτες. Θα πρέπει να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες και όχι να απομακρύνεται. Πρέπει οι νόμοι να είναι κατανοητοί και η διαδικασία νομοθεσίας να είναι και αυτή κατανοητή για τον απλό πολίτη στο όνομα του οποίου εμείς νομοθετούμε εδώ. Τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών καταδεικνύουν ότι οι πολίτες όλο και περισσότερο απομακρύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα για μια ακόμα φορά να χαιρετήσω το έργο που έκανε ο κύριος Καρίμ και να τον επενέσω για την προσπάθεια που έκανε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό της απόστασης των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζω λοιπόν την έκθεση Καρίν, θα την υπερψηφίσω και έχω μονάχα να θέσω ένα μικρό ερώτημα το οποίο ουσιαστικά έχει ξεπεραστεί που ήταν η δυνατότητα να διευρυνθεί ο χρόνος που δίνεται στα εθνικά κοινοβούλια για να εκφράσουν γνώμη για τα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 8 εβδομάδες να περάσει σε 12 εβδομάδες. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι εκθέσεις αυτές να αντιμετωπίζονται πιο ενδελεχώς από τα εθνικά κοινοβούλια και αυτό θα ενισχύσει και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα ήθελα να πω ότι αυτή η δυνατότητα δεν προβλέπεται από τις συνθήκες, αλλά αν το εγκρίνουν ομόφωνα το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό στο μέλλον μπορεί να έρθει και μέσα στη συνθήκη. Η κυρία Λόπες Μπερμέχο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, για πάρα πολλούς Ευρωπαίους υπάρχει άγνοια του γεγονότος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ε, προτείνει τους ευρωπαϊκούς ε, νόμους. Αυτό έγινε για να μην μπορεί να υπάρχει έκφραση των εργαζομένων ανθρώπων στην Ευρώπη και να μπορούν να περνούν μέσα στο κοινοβούλιο την άποψή τους. Το κάνει αυτό η Κομισιόν. Και μετά πέρα από το κοινοβούλιο θα πρέπει και οι κυβερνήσεις να εγκρίνουν τα νομοθετήματα αυτά και το πράττουν θέλοντας να προωθήσουν την απορριθμιστική και νεοφιλελεύθερη λογική της Ευρώπης. Η πολυπλοκότητα και η έλλειψη διαφάνειας σε αυτόν τον τρόπο νομοθέτησης βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης σήμερα. Υποτίθεται ότι τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας και της ε, επικουρικότητας και θα έπρεπε να οδηγούν σε μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία αυτή. Στην πράξη όμως είναι αρχές ασαφείς, όπως και εσείς οι συνάδελφοι το τονίζετε, οι οποίες εφαρμόζονται και ερμηνεύονται κατά το δοκούν πιστεύω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το βασικό πρόβλημα είναι διαφορετικό. Ο νέο φιλελευθερισμός. Μιλάει ο κύριος Καρίν για την επικουρικότητα και το να μπορούν τα εθνικά κοινοβούλια να αποφασίσουν για τις πολιτικές τους. Αλλά όταν μιλάμε για χώρες όπου υπήρξε ε, παρέμβαση της Τρόικα, όλα αυτά τα ξεχνάμε. Η αναλογικότητα επίσης αναφέρεται από εσά όπως και από την Κομισιόν με έναν τρόπο ο οποίο είναι πολιτικοποιημένο για να εμποδίσετε νέες νομοθετικές προτάσει, οι οποίες προσπαθούν να σταματήσουν τη διάβρωση των δικαιωμάτων εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λόπε, δέχεστε μία μπλε κάρτα από τη συνάδελφό σας την κυρία Άντερσον. Παρακαλώ. Να σας ευχαριστήσω για αυτήν την πρότασή σας. Βεβαίως και υπάρχουν κάποιες λύσεις που βρέθηκαν μέσω του ευρωπαϊκού εγχειρήματο, αλλά όχι αυτό εξαιτία της Τρόικα. Κοιτάξτε παραδείγματο χάρη τι έγινε με τους Ιρλανδούς. Μπορεί κανείς να πει ότι όλοι αυτοί που έχουν σταλεί εδώ για να εκπροσωπήσουν τους λαούς τους και όχι την Ευρωπαϊκή επιτροπή η οποία βεβαίω δεν έχει εκλεγεί από κανέναν Ευρωπαίο πολίτη. Συμφωνώ μαζί σα, κύριε Άντερσον, σε αυτή τη την τοποθέτηση. όντω. οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πραγματικά απογοητευμένοι λόγω των πολιτικών που ακολουθούνται από αυτό το κοινοβούλιο κατά των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Άντερσον, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή που αφορά την επικουρικότητα και την αναλογικότητα για το 2012 και 2013 περιέχει μια σειρά σωστών ορθών προτάσεων και μας οδηγεί προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τη δημοκρατική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς περιέχει όμως και μία σειρά μη ορθών προτάσεων, οι οποίες ε, παραδείγματο χάρη οδηγούν σε πολύ σημαντικές εκθέσεις αντικτύπου. Οι εκθέσεις αντικτύπου, η αξιολόγηση αντικτύπου δεν είναι κάτι το εύκολο, δεν είναι εύκολο να διεκπαιρεωθεί. Δηλαδή πρόκειται για αριθμούς οι οποίοι πολλές φορές δεν είναι ορθοί, δεν είναι αριθμοί, αξιόπιστοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιος να αποκτήσει αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά την προστιθέμενη κοινωνική αξία μιας πολιτικής ενός ε, νομοθετικού κειμένου. Ε, η αξιολόγηση λοιπόν, η έκθεση αντικτύπου είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να γίνει. Πρέπει να περάσει χρόνος. Δεν θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλές τέτοιες εκθέσεις αντικτύπου να είναι αποτελεσματική. Θέλουμε να γίνεται έλεγχος της επικουρικότητας βεβαίως στην πράξη. 15 από τα εθνικά κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν αυτόν τον μηχανισμό ελέγχου της ε, επικουρικότητας και λειτουργεί το σύστημα ελέγχου μέσω των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μία πράσινη κάρτα, έτσι όπως προτείνεται, σίγουρα είναι μία πάρα πολύ ε, καλή ιδέα. Θα πρέπει να την εξετάσουμε και ελπίζω ότι η επόμενη έκθεση θα είναι ακόμα καλύτερη. Ο κύριος Μπάτεν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση αυτή όσον αφορά την ευκαιρικότητα και την να αναφέρεται στο άρθρο 5 της ε, συνθήκης όσον αφορά την άσκηση μιας ε, αρμοδιότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που αυτή μπορεί να γίνει σε, μεγαλύτερο τρόπο, σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται ουσιαστικά για τον έλεγχο της δημοκρατικότητας ε, μιας πολιτικής. Αν δηλαδή μπορεί να γίνει με καλύτερο, πιο αποτελεσματικό τρόπο από τα εθνικά κοινοβούλια η δημιουργία ενός τέτοιου νομοθεσίας. Πριν από 20-25 χρόνια θυμάμαι ότι είχε προταθεί ένα βραβείο, ε, χρήματα μάλιστα, όταν χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο η επικουρικότητα και όταν η νομοθεσία γίνεται στο τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει ίσως να δούμε αν όλα αυτά για τα οποία νομοθετούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τους βραστήρες μέχρι θέματα, αλλά που αφορούν τελικά πολύ περισσότερο το τοπικό ή το εθνικό επίπεδο, γίνονται ορθά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια πράσινη, μια κίτρινη κάρτα που θα αφορά κάποια κράτη-μέλη, όχι ένα μεμονωμένο, αλλά 15 κράτη-μέλη, για να σταματήσει μια τέτοια νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ίσως μας εμποδίσει να έχουμε κάποιες γελίες καταστάσεις όπως αυτές που βλέπουμε στο YouTube έναν υπουργό ο οποίος περιγράφει αυτή την κατάσταση, ο David Cameron δίπλα του γελάει χασκογελάει. Βλέπετε λοιπόν ότι βεβαίως η αναλογικότητα είναι πολύ σημαντική, η επικοινωνικότητα εξίσου και ίσως αυτές οι σκέψεις που κάνουμε σήμερα θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο ερώτημα γιατί οι Βρετανοί σήμερα κινδυνεύουν τις 23 Ιουνίου να ψηφίσουν για να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λεμπρετό για δύο λεπτά, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η διαδικασία της ε, κίτρινης κάρτας είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να υποχρεώσουν την Κομισιόν να δεχτεί και να εφαρμόσει την αρχή της επικουρικότητας. Υποχρεώνει την Κομισιόν να επανεξετάσει μια νομοθετική πρόταση αν αυτή έχει σταθεί αντικείμενο διαμαρτυριών αιτιολογισμένης γνώμης από το 1 τρίτο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η διαδικασία όμως αυτή της κίτρινης κάρτας μόνο μια φορά ανάγκασε και έψε την Κομισιόν να εγκαταλείψει μια πρόταση το 2012 για την πρόταση Μόντι 2 που έθετε ένα το δικαίωμα της απεργίας. Είναι πολύ ισχνό αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα γιατί σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η Κομισιόν αντιμετωπίζει με αλαζονία τις κίτρινες κάρτες. Είναι λοιπόν μια απάτη η ιστορία της ε, κίτρινες κάρτας. Η Κομισιόν μπορεί να τα παρακάμπτει με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις που χρησιμοποιεί κατά κόρον όταν τη βολεύει. Η κατάσταση αυτή λοιπόν δεν μπορεί να διορθωθεί με το να έχουμε μια έκθεση που ζητά από την Κομισιόν να έρθει σε διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και να βελτιώσει τι εκθέσει αντικτύπου. Προτείνει βέβαια να υπάρξει αυτή η διαδικασία πράσινη κάρτα που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να δίνουν προτάσει στην Κομισιόν. Αυτό όμως θα θυμίζει τις αιτήσει που έδιναν στο βασιλιά ή και τευτικά οι πολίτες στο καθεστώς της Γαλλίας όταν ήταν ακόμα βασιλεία. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα δεν πηγαίνουμε πουθενά. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πραγματική διαδικασία κόκκινη κάρτα που επιτρέπει σε οποιοδήποτε κράτο μέλο να αντιταχθεί σε μια πρόταση τη Κομισιόν όταν θεωρεί ότι θίγονται τα εξωτικά συμφέροντά του. Η κόκκινη αυτή κάρτα θα είναι δικαίωμα βέτο που επιτρέψει σε κάθε κράτος να εξασφαλίσει το σεβασμό της κυριαρχικότητάς του. Θα είναι ένα πρώτο λοιπόν βήμα προς μια Ευρώπη εθνών που είναι ακριβώς αυτό το οποίο εγώ προσωπικά εύχομαι. Ευχαριστώ. Κύριος Συναγνός, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δυσπιστία και ο ευρωσκεπτικισμός των πολιτών είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης προς τις αρχές της αναλογικότητας και επικουρικότητας στη χάραξη ενωσιακών πολιτικών προφανώ δεν φταίνε οι λαοί τη ευρώπη όση προπαγάνδα και αν χρησιμοποιείται. παράδειγμα η ελλάδα. ο ελληνικό λαό δεν είναι τεμπέλης διεφθαρμένο και άτιμο μόνο ευκολόπιστο και παραπλανημένο από πολιτικού αλτιμπάγκου και κατευθυνόμενα μέσα μαζική ενημερώσεω εγχώρια και ξένα. έξι χρόνια τον παραπλανούν ότι τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί νόμοι επιβάλλονται προ όφελό του και με γνώμονα τη βιωσιμότητα τη πατρίδος του ενώ οι ίδιοι τηρούν υπέρογκου τραπεζικού λογαριασμού και εξωχώρε εταιρείε σκάνδαλα που καλύπτονται λίστες με φορολογικές ατασταλίες που ποτέ δεν διερευνούνται επίουργοι πολιτικοί που κρύβονται πίσω από τις κοινοβουλευτικές ασυλίες. αλήθεια πόσο αναλογικό και επικουρικό είναι αυτό προς τους πολίτες που δεν έχουν να φάνε ή να πληρώσουν τα φάρμακά τους. καμία πολιτική μνημονίου και κανένας εφαρμοστικός νόμος δεν τήρησε τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας για τους έλληνες μόνο τις αρχές της τιμωρίας της τραπεζικής μακροοικονομίας και του πλιάτσικου στην ιδιωτική ακίνητη και κινητή περιουσία τα ψέματα πλέον τελειώσαν και μαζί τελειώνουν και οι αποτυχημένες δεξιές και αριστερές κυβερνήσεις. εμείς σαν εθνικιστές λέμε ναι στην ευρώπη των λαών και των εθνών με δικαιοσύνη όμως στην αναλογικότητα και επικουρικότητα. ευχαριστώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Επιτροπές ε, Νομικών Θεμάτων για την υποστήριξη αυτής της έκθεσης και ιδιαίτερα τον κύριο Καρίμ για το γεγονό ότι δέχτηκε συμβαστικέ λύσεις. Για μένα το θέμα τη αναλογικότητα και τη επικουρικότητα είναι από τα κυριότερα θέματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε στη διαδικασία νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα πρέπει να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ώστε να υπάρξει μια καλύτερη σχέση μεταξύ εθνικών κρατών και, και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η εφαρμογή αυτή της διαδικασίας δεν πρέπει να είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να επηρεάσουν αυτή τη διαδικασία. Στο Συμβούλιο των Υπουργών βρίσκονται υπουργοί οι οποίοι είναι υπόλογοι έναντι των εθνικών του κοινοβουλίων. Αυτή η αρχή λοιπόν ε, είναι απαραίτητο να μπορέσει να λάβει σάρκα και όστά. Αυτό ζητούν οι πολίτες μας. Δεν πρέπει λοιπόν αυτή η αρχή να γίνεται υπό τη μορφή εποπτείας και ελέγχου, αλλά θα πρέπει να είναι και μια βάση για τις κοινέ ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Δεν θα είναι. Δεν πρέπει να είναι για να μπλοκάρει πρωτοβουλίες, αλλά για να ενισχύει πρωτοβουλίες. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η έκθεση θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένες ενέργειες και προτάσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοφεράτη έχει το λόγο. Ένα μισό λεπτό. Κύριε Επίτροπε, όπως γνωρίζετε, η αρχή αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές και πολύ ευαίσθητες. Όχι μόνο δύσκολες στο να υλοποιηθούν, αλλά και στο να εξισορροπήσουν ε, να με, ε, μεταξύ τους. Πολλοί συνάδελφοι δεν το υπογράμμισαν αυτό και όχι τυχαία. Ποιο είναι το, τα πορίσματα αυτής της έκθεσης, ότι όλες οι ε, μεταγενέστερες μορφές ελέγχου τελικά καταλήγουν στο να αφαιρέσουν τη διαφάνεια από τις διαδικασίες και επιπλέον αντιστρέφουν αυτό που για μας είναι μια θετική διαδικασία, δηλαδή να δώσουμε περισσότερη αυτονομία και εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, επανερχόμαστε στο να αναθέτουμε ευθύνες που δεν είναι απαραίτητο αυτό προς τα κρατημέλη. Δηλαδή, πρόκειται στην ουσία για μια διάταξη που μας απομακρύνει από τους στόχους που εδώ εμείς ε, ε, για τους, μάλλον που εδώ εμείς αντιπροσωπεύουμε και που, για τους οποίους μας εξέλεξαν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ε, εδώ θέλω να τονίσω ότι έχουμε, βρισκόμαστε ενώπιον μια υποθετική λύση σε αντίθεση με άλλε διατάξει που είναι υποσυζήτηση αυτές μάλιστα τι ημέρε, γιατί θα αντιμετωπίσουμε και θα ψηφίσουμε αύριο γι' αυτό. Δεν είναι αυτό συνεπή με τη Διοργανική Συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία και επίση έρχονται σε αντίθεση με τις συμβιβαστικέ που θα ψηφίσουμε για την ΡΕΦΙΤ. Δηλαδή αυτή η κατεύθυνση θα πρέπει αμέσως να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα, ενάμιση λεπτό ο κύριος Λούκε. Ένα λεπτό έχω εγώ για σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση. Η επικουρικότητα, η αναλογικότητα είναι δύο βασικές αξίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όμως να χρησιμοποιούνται στην πράξη κατά τη διάρκεια της νομοθετικής μας εργασίας και να μην τις παραβιάζουμε. Αυτό που βλέπουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ε, πρόταση για την ε, ουσιαστική στήριξη της, ε, του τρίτου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης και βεβαίως το θέμα της θεσμικής εγγύησης για τις διαφορετικές δραστηριότητες των τραπεζών, αποταμίευση από την άλλη, επενδύσεις και τους μεγάλους κινδύνους οι οποίοι σήμερα δεν αντιμετωπίζονται από τα οικονομικά μέτρα. Βλέπουμε ότι κάτι λάθος εδώ έχει γίνει. Είναι αντίθετο από την αρχή της επικουρικότητας αυτό που προτείνεται για την Τραπεζική Ένωση και για τα πρόσφατα μέτρα για τη διασφάλιση των εγγύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπιλμπάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιχωρικότητα και αναλογικότητα. Αυτά είναι βασικά στοιχεία δομικά για μια αρμονική οικοδόμηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μηχανισμοί που έχουν θεσπιστεί αυτή τη στιγμή για να είναι σεβαστέ αυτέ οι αρχέ είναι φορμαλιστικέ και ανεπαρκεί και δεν επιτρέπουν στι ε, περιοχέ ε, τη ε, Ευρώπη που έχουν νομοθετικέ αρμοδιότητε να χρησιμοποιήσουν αυτέ τι διαδικασίε. Παραδείγματο χάρη στη δική μου χώρα η διαδικασία αυτή αν δεν συμφωνούν οι αυτόνομες περιοχές με την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, δεν περιλαμβάνεται και η γνώμη τους σε αυτά τα οποία λέει το κοινοβούλιο. Επομένως, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι για την νομοθεσία που μας επηρεάζει. Όλα αυτά απομακρύνουν περισσότερο τον πολίτη και θίγουν τη συμμετοχή των πολιτών μας. Μας έχει δείξει η πείρα ότι πρέπει να τροποποιηθεί αυτή η διαδικασία και όπως λέει η έκθεση του κ. Κάρεμ. Δεν αρκεί ο έλεγχος εκ των προτέρων είναι απαραίτητο να γίνεται και μία εκ των υστέρων έκθεση για την εφαρμογή και τη λειτουργία των ε, ευρωπαϊκών οδηγιών υπό το πρίσμα της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Πρέπει να τα πάρουμε όλα αυτά λοιπόν σοβαρά αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια ομοσπονδιακή Ευρώπη και μια πραγματική ένωση. Δηλαδή μια ένωση θεληματική όλων των μελών που την απαρτίζουμε. Πρέπει λοιπόν να μην γίνεται αυτό το οποίο γίνεται τώρα, όπου μονάχα οι δεσμοί μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους. Η Λάουρα Φεράρα για ένα λεπτό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε στην εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας όταν σωστά ερμηνεύεται σημαίνει ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σε ένα επίπεδο όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Αυτό είναι πολύ θεμελιώδης σημασία για το κίνημα των πέντε αστέρων. Δεν πρόκειται για ένα μέσο άμεσης δημοκρατίας, αλλά σίγουρα πρόκειται για μια αρχή που στόχο έχει να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες της, εγγυόμενη την σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών μελών και τη δράση σε τοπικό επίπεδο ο κάθε φορά που αυτό είναι απαραίτητο. Ε, περιμένουμε λοιπόν, την εκφράζουμε μάλλον την εκτίμησή μας για αυτή την έκθεση, γιατί περιγράφεται την αρχαία αυτή, αλλά και τους περιορισμούς στη σωστή της ερμηνείας. Υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα την παράγραφο 29 της έκθεσης, τη στιγμή όπου η συμμόρφωση με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας ε, συζητώνται, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει πιο αποτελεσματική και εξωκρατική την ε, κατάσταση κατάσταση στις διαδικασίες, στις γραφειοκρατικά περίπλοκες όπου διαπιστώνονται σε ε, περιστατικά διαφθοράς και θα πρέπει επίσης η επικουρικότητα να χρησιμοποιείται και να λαμβάνεται υπόψη και στο πλαίσιο των διαφόρων εμπορικών, διεθνών εμπορικών συμφωνιών που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Um, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήταν πολύ καλύτερα αν μιλούσατε λίγο πιο αργά. Για όλους θα ήταν πολύ καλύτερα, ώστε να μπορούν καλύτερα οι διερμηνείς να σας μεταφράσουν. Αν στις δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Υπήρξε το δημοψήφισμα στην Ολλανδία. Τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας εκφράστηκαν κατά ενός ε, μέτρου ευρωπαϊκού που αντίκειται στην αρχή της επικουρικότητας. Κανονικά η αρχή της επικουρικότητας θα έπρεπε να εμποδίσει αυτήν την ε, ένα η επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρμοδιότητες οι οποίες σε κανένα ε, τομέα δεν θα έπρεπε να ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαβάζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δεν πρόκειται για τις αποκλειστικές της αρμοδιότητες μπορεί να παρέμβει αποκλειστικά και μόνο, διαβάζω το κείμενο, παραθέτω, οι στόχοι δεν μπορούν να ρυθμιστούν, να επιτευχθούν σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, αλλά μόνο εάν αυτοί οι στόχοι δεν μπορεί παρά να υλοποιηθούν καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό όμως είναι ένα πάρα πολύ ασαφές κείμενο. Οι υπέρμαχοι της περαιτέρω διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να υποστηρίξουν ότι αυτή η φράση αυτό σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες θα πρέπει να συνδυάζονται πάντα σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι αν μια απόφαση λαμβάνεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το ευρωπαϊκό η επικουρικότητα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αποτελεσματική. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτοί που υποστήριζουν μια τέτοια ερμηνεία δίνουν λευκή επιταγή σε αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν την Ευρώπη Ομοσπονδία. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε κάτι τέτοιο. Αν κάτι τέτοιο είναι η κατεύθυνση που επιλέγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να περάσουν οι ευρωπαϊκές χώρες από δημοψηφίσματα. Κάτι που σίγουρα θα δημιουργήσει αναταράξεις σε μια τέτοια ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Αυτή η φράση λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνεύεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Για μένα δεν έχει απολύτως καμία βαρύτητα. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Ζαμπόρσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Καρίμ, για το κείμενο που μας έχει υποβάλει. Πολλά εθνικά κοινοβούλια συμφωνούν με αυτές τις προτάξεις. Πρέπει να ενισχύσουμε τον δημοκρατικό, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα πρέπει σίγουρα να πλησιάσει η Ευρώπη τους Ευρωπαίους πολίτες. Και κάθε φορά που ρωτούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες απαντούν προς αυτή την κατεύθυνση. Το ψήφισμα αναφέρει σαφέστατα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα κόστος και δεν μπορεί οι ανησυχίες, οι επιφυλάξεις των Εθνικών Κοινοβουλίων, οι πρωτοβουλίες των πολιτών που εκφράζουν αυτές τις ανησυχίες να αγνοούνται παντελώς από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ξέρετε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες που υπέβαλαν αυτό το ψήφισμα δεν γνωρίζουν την αρχή της επικουρικότητας ούτε της αναλογικότητας. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση πριν ψηφίζεται ένα κείμενο εδώ στην Ολομέλεια, να ελέγχεται κατά πόσο έχει τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Θα πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά αυτές τις έννοιες, αλλιώς η οργή των πολιτών θα οδηγήσει στην κατάρρευση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό. Η Μερσέντες Μπρέσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω πως η συζήτηση για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα χαρακτηρίζεται και από τους τόσους ευρωσκεπτικιστές που μας λένε πως η Ευρώπη δεν σέβεται αυτή την αρχή. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν δει κανεί τον πολύ περιορισμένο αριθμό κίτρινων καρτών και πορτοκαλί καρτών που όχι μόνο φτάνουν μέχρι τέλος αλλά και το πολύ περιορισμένο αριθμό των όσων ξεκινούν τη διαδικασία, γιατί για να ξεκινήσει μια διαδικασία παράβασης της επικουρικότητας ε, θα πρέπει κανείς να αποδείξει την, την παράβαση. Αυτό μας δείχνει λοιπόν, επειδή συμβαίνει αυτό πολύ σπάνια, πως η παράβαση γίνεται από πλευράς ε, της ε, Κομισιόν και είναι δύσκολο να αποδείξει κανείς την ύπαρξη παράβασης. Εγώ πιστεύω λοιπόν πως αυτή η έκθεση έχει σε μεγάλο βαθμό επηρεαστεί από αυτήν την ε, παρατήρηση και κινδυνεύει να επιβαρύνει και να ζημιώσει την άλλη σημαντική αρχή που είναι η αρχή της απλοποίησης και της καλύτερης νομοθεσίας ή να παρατείνει επαόριστο την ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ε, γι' αυτό και πιστεύω πως κάποια στοιχεία δεν θα πρέπει να ψηφιστούν κάτι τώρα ακόμα για την πράσινη κάρτα. Είναι ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά θα πρέπει να ενταχθεί σε μία ε, συνθήκη και να μην χρησιμοποιηθεί και να αποτεθεί σε εφαρμογή τώρα, γιατί θα πρέπει να συνδέεται με την ε, ε, νομοθετική πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Μόνο με αυτό θα πρέπει να συνδεθεί. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριος Μαριάς. Κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται στην ένωση με τις συνθήκες ανήκει στα κράτη μέλη. με τη ρύθμιση αυτή καθορίζεται πανηγυρικά ότι το τεκμήριο αρμοδιότητας ανήκει στα κράτη μέλη τα οποία διατηρούν τα αποκλειστικά κυριαρχικά τους δικαιώματα σε όλα τα πεδία πλην εκείνων στα οποία η συνθήκη με βάση την αρχή της δοτής αρμοδιότητας απονέμει εξουσία δράσης στα όργανα της ευρωπαϊκής ένωσης τα οποία μάλιστα όταν δρουν στο πεδίο των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων οφείλουν να σέβονται τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. στην ελλάδα η ευρωπαϊκή επιτροπή και η τρόικα και η εκουτού παραβιάζουν συνεχώς βάναυσα την αρχή της δοτής αρμοδιότητας καθώς δρώντας σε πεδία που δεν ανήκουν καν στις αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής ένωσης επιβάλλουν μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις αυξάνουν τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας διαλύουν το ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις και απαιτούν ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας κύριοι της κομισιόν σταματήστε επιτέλους να παρανομείτε και να παραβιάζετε τις συνθήκες της ευρωπαϊκής ένωσης. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Έχει το λόγο η κυρία Εστάρας Φεραγκούτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον Ασχητή για αυτή την έκθεση και όντως οι αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας είναι σε για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το σημείο κίνησης των ευρωπαϊκών πολιτικών γιατί ε, αυτή η πολιτική επικουρικότητα φέρνει πιο κοντά τον πολίτη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια για να νομοθετήσει το ίδιο και η αρχή της αναλογικότητας. Γι' αυτό και είναι σωστό και έχει νόημα ε, να οποιαδήποτε δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσαρμόζεται στον ε, στόχο που επιδιώκει. Είναι σημαντική η έκθεση αυτή γιατί στόχος είναι να εγγυηθούμε την αποτελεσματικότητα και την ε, δημοκρατική νομιμότητα στην λήψη αποφάσεων. Και πάντως ε, ενισχύεται έτσι το ευρωπαϊκό σχέδιο. Μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουν φτιαχτεί μια ολόκληρη σειρά από κάρτες από πλευράς των εθνικών κοινοβουλίων ώστε να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί για να μπορεί σωστά να ελέγχεται η εφαρμογή αυτή τη αρχή αυτών των αρχών, τη επικροτικότητα και τη αναλογικότητα. Αυτή η διαδικασία γίνεται φυσιολογικά, ωστόσο είναι αλήθεια πώ όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να είναι ε, ευέλικτοι να είναι λογική και απλή και αποτελεσματική. Το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις διοικητικές, τους διοικητικούς μηχανισμούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς καθώς και το να ενισχυθούν αυτές οι αρχές. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η Εύλην Ρέγνερ για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η επικορικότητα θα έπρεπε να σημαίνει να είμαστε πιο κοντά στους πολίτες, να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Η, η επικουρικότητα όμως δεν σημαίνει αδράνεια και αδυναμία δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην νομοθεσία. Οι άνθρωποι στην Ευρώπη πραγματικά θέτουν αυτό το ερώτημα. Πώς λειτουργεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι τόσο πολύπλοκες οι διαδικασίες της. Και όσο πιο πολύ βλέπουμε τα πράγματα αυτά, είναι όλο και πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Αυτό οδηγεί σε ένα κικαιώνα μέσα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιες είναι οι αρμοδιότητες του καθενός, αντί να έχουμε πραγματικά καθορισμένες αρμοδιότητες και να ασκούν τα Εθνικά Κοινοβούλια το δικαίωμα του ελέγχου επικυρικότητας, όπως έχουν το δικαίωμα. Το να υποστηρίξουμε κάτι είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά το να εμποδίζουμε είναι κάτι το οποίο πάντα δημιουργεί προβλήματα. Εδώ αναφέρεται ότι στην έκθεση ότι και ο ίδιος ο έλεγχος επικουρικότητας πολλές φορές δεν λειτουργεί και γι' αυτό προτείνει και τη χρήση μιας πράσινης κάρτας και όχι μονάχα να χρησιμοποιείται η κόκκινη κάρτα η οποία μπορεί να σαμποτάρει θετικές πρωτοβουλίες όπως παραδείγματος χάρη θέματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό διάλογο. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι δεν πρέπει η διαδικασία αυτή επικουρικότητας να οδηγήσει και σε αποδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου και των κοινωνικών εταίρων. Και θέλω να τονίσω ότι υπήρξαν και πολύ καλύτερες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για την επικουρικότητα ώστε να εφαρμοστεί με πιο καλό τρόπο η αρχή της επικουρικότητας σεβόμενη και τα δικαιώματα των κοινωνικών εταίρων. Ευχαριστώ κυρία Ρέγνερ. Ενάμιση λεπτό κυρία Κολοβόσκα Ραβέσκα, Κάπως έτσι. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε. Να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή για αυτή την εξαιρετική του έκθεση που ουσιαστικά υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερη επικουρικότητα ενώ Φυσικά συνεχίζεται η διαδικασία η νομοθετική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καλύτερη και περισσότερη συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων στην νομοθεσία την ευρωπαϊκή. Λιγότερη γραφειοκρατία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στα κράτη-μέλη, στα Εθνικά Κοινοβούλια, η Κίτρινη Κάρτα, η Πράσινη Κάρτα, όλες αυτές οι προτάσεις θα βοηθήσουν να σταματήσει κάποια νομοθεσία, να εμποδιστεί είτε να συνεισφέρουν τα κράτη-μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια στη δημιουργία νέων νομοθετικών προτάσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε περί τίνος πρόκειται. Τι είναι ακριβώς αυτή η επικουρικότητα. Πρόκειται για έναν από τους ακρογωνιαίους λήθους της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Σε επίπεδο κρατών θα πρέπει να γίνονται οι περισσότερες προτάσεις και να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο αυτό που μπορεί να γίνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να μην ξεχνάμε την επικουρικότητα λοιπόν, γιατί παραβιάζοντας αυτές τις αρχές δημιουργούμε αντιπαραγωγικά μέτρα και εμπόδια για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κάφμαν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η άποψή μου είναι ότι τα τελευταία έξι χρόνια δείξαμε ότι το σύστημα αυτό βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας και η αρχή της επικουρικότητας λειτουργήσαν ικανοποιητικά. Ουσιαστικά επιστήσαμε την προσοχή όλων μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών στην αρχή της επικουρικότητας και αποδείχθηκε ότι υπάρχει κατανομή αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα. Και αυτό είναι κάτι πολύ ε, θετικό για την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας που λαμβάνει υπόψη του την ε, επικουρικότητα. Και αυτό για να υπάρξει σεβασμός των αρμοδιοτήτων ε, του ευρωπαϊκού επίπεδου, του εθνικού επίπεδου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όλοι επιθυμούμε να υπάρξει καλύτερη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, καλύτερη νομοθεσμία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα σύστημα με πολλά επίπεδα, ένα περίπλοκο σύστημα και θα πρέπει να είναι σαφές για να μπορέσουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες να κατανοήσουν το τι συμβαίνει, ποιος είναι αρμόδιος γιατί, ποια είναι ακριβώς αυτή η κατανομή αρμοδιοτήτων που δεν θα πρέπει να οδηγεί σε σύγχυση. Βλέπετε τι έγινε παραδείγματος χάρη με τις κάτω χώρες, με το δημοψήφισμα στην Ολλανδία οι ηγέτες κάποιων λαϊκιστικών και δημαγωγικών κομμάτων έχουν πολλές φορές ε, δημιουργήσει, όπως και σε άλλες χώρες, τρευλώσεις, δημιουργώντας μια εικόνα της κακής Ευρώπης και αντίθετα παρουσιάζοντας το τοπικό ή εθνικό επίπεδο σαν το καλό. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε τέτοια στρέβλωση της εικόνας της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να ενισχυθούν και από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια και τα περιφερειακά κοινοβούλια να συνεργαστούν για καλύτερη νομοθεσία. Ο κύριος Μπούντα για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία του. Ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια ε, ασχολήθηκαν με τον εντοπισμό απαραίτητων ε, μηχανισμών για την υιοθεσία νομοθεσία που αντιστοιχεί ταυτόχρονα στι διεθνεί απαιτήσει αλλά και στην ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η σεβασμός των αρκών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας μέσα στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας βλέπουμε ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η ανάγκη των των Ευρωπαίων πολιτών να, γίνεται σεβαστές αυτές οι δύο αρχές στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ε, και να προταθούν, ε, να προτείνονται μάλλον προβλήματα, μάλλον λύσεις στα προβλήματα που εντοπίζονται, ε, ξεκινώντας από την αρχή πως αυτές οι δύο ε, ε, αυτά τα δύο σημεία κίνηση τη Ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει λεπτομερώς να ελέγξει κατά πόσο γίνονται σε σεβαστές αυτές οι αρχές. Ωστόσο, ε, θέλω να υποβάλω κάποιους προβληματισμούς. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως οι μελέτες αξιολόγηση έχουν στόχο μόνο τα αρχικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας ενώ οι νομοθετικές προτάσεις μπορεί να έχουν να, να, να υποστούν διάφορες τροπολογίες ε, τροποποιήσεις στη διάρκεια της έγκρισης γι' αυτό για να σεβαστούμε το συμφέρον των πολιτών ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια ο κύριος Πόσπισιλ για 1,5 λεπτό Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε και εγώ θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έκθεση αυτή Εγώ υπήρξα αρμόδιος για τα θέματα εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας και θέλω να τονίσω ότι υπήρξαν κάποιες προτάσεις οι οποίες έγιναν τότε δεκτές, αλλά υπάρχουν πολλές οδηγίες στις οποίες δεν υπάρχει πραγματική εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και της ε, αναλογικότητας πέραν καθαρά τυπικών διατυπώσεων. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια σοφή, σωστή αντιμετώπιση για τις ε, προτάσεις αυτές, γιατί πολλές φορές αναφέρεται το θέμα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας μόνο σε τυπικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο λοιπόν η Κομισιόν να σέβεται περισσότερο τα δύο αυτά κριτήρια στην νομοθεσία και να μπορεί αποτελεσματικά να αξιολογεί την λειτουργία και το σεβασμό αυτών των αρχών. Είναι επίσης σημαντικό να λάβουμε υπόψη και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να σκεφτούμε όλοι ότι είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη περισσότερο η άποψη των εθνικών κοινοβουλίων και τις περιπτώσεις που έχει υπάρξει μια κίτρινη κάρτα, μια διαδικασία κίτρινης κάρτας, νομίζω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να δίνει περισσότερη προσοχή στα θέματα αυτά και νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σεβασμό για τι κίτρινε κάρτε. Ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Νεγκρέσκου για ένα λεπτό. principiile solidarității subsidiarității și proporționalității sunt importante. ele au fost create. οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας είναι σημαντικές για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ισορροπία των εξουσιών αλλά είναι και ο τρόπος για να μπορούν να υποβάλλονται σωστότερα νομικά κείμενα. Όμως δεν συμφωνώ με τον εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργηθεί για να διατηρηθεί η ειρήνη, για να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, για να τηρούνται οι κοινοί κανόνες, για να αναπτυχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εισηγητή έλεσε ότι δεν θα πρέπει να φοβόμαστε, να φοβόμαστε την Ευρώπη και δεν την φοβάμαι, αλλά, φοβ, αλλά εσείς τη φοβάστε. Γιατί εδώ ακούγονται διάφορες φωνές. Εγώ υποστηρίζω την ιδέα για την έκφραση της γνώμης ε, του τοπικού επίπεδου και του εθνικού επίπεδου. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνεται με βάση υπάρχοντες μηχανισμούς και με ισορροπημένη σχέση και όχι με λαϊκίστικα μηνύματα. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό, Ιβαν Γιάκοφτσίτσε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάθε πολιτική είναι τοπική πολιτική, διότι κάθε πολιτική συμπεριλαμβανομένων των δικών μας που εγκρίνουμε εδώ αντικατοπτρίζονται και επηρεάζουν και το τοπικό επίπεδο. Επηρεάζουν τους πολίτες μας που ζουν σε συγκεκριμένη κοινότητα, πόλη ή περιφέρεια. Γι' αυτό τελικά όλες οι πολιτικές είναι τοπικές και γι' αυτό και πιστεύω ότι η αρχή της επικουρικότητας είναι εξαιρετικά σημαντική ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνεται καλύτερα κατανοητή από τους πολίτες διότι πρέπει να παραδεχτούμε πως υπάρχει πρόβλημα με την ταυτότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών προφανώς προφανώς δεν μπορούν ε, όλες οι πολιτικές να ασκούνται σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να υπάρχουν πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα πρέπει να μεταφράζονται και να ευθυγραμμίζονται σε τοπικό επίπεδο. Και έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα περνάμε στην ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Επίτροπο Γιώργοβα. Έχετε το λόγο. thank you very much for... Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα σχόλια και τις ερωτήσεις σε αυτό το σημαντικό θέμα. Θα ήθελα με την ευκαιρία να επαναλάβω αυτό που ανέφερε ο κύριος κύριος με την πρόταση για τον Ευρωπαίο Συγγελέα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικότερα και η Ένεση. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, αιτήματα ενημέρωση από Εθνικά Κοινοβούλια. Έχω ήδη πει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισκεφθεί σε 270 τουλάχιστον ε, περιστάσεις Εθνικά Κοινοβούλια, εκ των οποίων περιστάσεων οι 10 τουλάχιστον της δικής μου, ήταν δική μου επίσκεψη ε, και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να πηγαίνουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια για να εξηγούμε πώς τροποποιήθηκε η πρόταση από αποκεντρωμένη, αποκεντρική σε αποκεντρωμένη δομή και πιστεύω ότι τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να δουν ένα σαφές ενδιαφέρον εξήγηση και τοποθέτηση σε σχέση με την επικουρικότητα από την ε, πλευρά μας. Αυτός είναι ε, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση νομίζω το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν αντικαθίστανται τα εθνικά εισαγγελικά όργανα, αλλά ενισχύονται με τον θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Αυτό για άλλη μια φορά ένα παράδειγμα του πώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε και την επικοινωνία με τα εθνικά κοινοβούλια. Και να ενισχύσουμε γενικά την επικοινωνία. Οι υπηρεσίε μα είναι στη διάθεσή σα για την συζήτηση πτυχών επικουρικότητα και αναλογικότητα στι προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλου του βουλευτέ για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο εισηγητή για δύο λεπτά. Κύριε Σκαρίμου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα μας ανέφερε και που κατέγραψε και την τεράστια στήριξη της οποίας έτυχαν ε, οι ιδέες μου κυρίως από τον ε, κύριο Τίμερμανς. Και αυτό το βρίσκεται στο πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν. Όμω ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες που συμμετείχαν στην ε, συζήτηση σήμερα για να προαγάγουμε με επικοδομητικό πνεύμα αυτέ μα τι παρατηρήσει. Παρότι στις περιπτώσεις των περιπτώσεων υπάρχουν διαφωνίες οι προτάσει του βασίζονται σε ένα επικοδομητικό πνεύμα και μια θετική ανάλυση για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους. Ένα-δύο ζητήματα που θα ήθελα να θίξω εν συντομία. Πρώτον, σε σχέση με την κόκκινη κάρτα, δεν πρόκειται για βέτο. Ποτέ δεν είχε προταθεί ως βέτο, ούτε υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός. Όμως, ποιο είναι το ζήτημα. Αν έχουμε τα υπόλοιπα μέτρα που ε, φέρνουν τα εθνικά κοινοβούλια πολύ πιο κοντά στη δική μας ε, διαδικασία υιοθέτηση και λήψη αποφάσεων, ποτέ δεν θα, θα βρεθούμε σε αυτή την περίπτωση που το Κοινοβούλιο θα ε, προχωρήσει στην κόκκινη κάρτα, πόσο μάλλον σε δικαίωμα κυρία. Για την εμπορικότητα που ανέφεραν οι συνάδελφοι, πρέπει να το εξετάσουμε και μέσω πρόθεσμα και στο τέλος. Όμως αυτές οι αξιολογήσεις δεν είναι δεσμευτικές αποτελούν μια μέτρηση για να διασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε αποκλίνει πάρα πολύ από την αρχή της επικουρικότητας και ότι γίνεται η δουλειά στο επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να γίνεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παράταση της αρχικής ε, περίοδου των 8 εβδομάδων, συμφωνώ ότι θα πρέπει όλα αυτά να ενσωματωθούν στις συνθήκες κατά την επόμενη επικαιροποίησή τους. Και τέλος, από την πλευρά της άκρας δεξιάς ε, είχαμε αρκετά σχόλια αρκετά ενδιαφέροντα για μένα, ιδίως από τους εκπροσώπους του UKIP που δεν είναι πλέον εδώ. Είπαν λοιπόν, πολλά είπαν, αλλά σε ό,τι αφορά τα τεχνικά ζητήματα έκαναν δύο παρατηρήσεις που ήταν και οι δύο απολύτως λανθασμένες. Ε, περιέγραψαν την κόκκινη κάρτα ως κίτρινη κάρτα. Και είμαι σίγουρος ότι και ο Βρετανικός λαός θα τους δείξει την κόκκινη κάρτα πολύ γρήγορα. Και είναι το 13% και όχι η πλειοψηφία, θα έλεγαν εκείνοι. Κόκκινη κάρτα λοιπόν στις 3 Ιουνίου. Ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνει τη συζήτηση για την έκθεση αυτή.